Bonjour. Euh. Καλησπέρα, καλημέρα σας. Σας καλωσορίζω θερμά σε αυτή την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ανάπτυξης μετά τις θερινές διακοπές. Το καλοκαίρι που μας πέρασε ήταν πολύ πλούσιο σε θέματα που μας ενδιαφέρουν και κυρίως της ανθρωπιστικής βοήθειας θα συζητήσουμε αυτό το θέμα και της Συρίας και της ε, Κεντρικής Αφρικής προς το τέλος της συνεδρίας. Ξεκινάμε ως ήθιστε με την έγκριση της σας διάταξης. Η κυρία Κρέτσου μας ζήτησε να διαγράψουμε το σημείο που είχε προβλεφθεί για το απόγευμα στις 3.30 την έκθεσή της δηλαδή για τις τοπικές αρχές και την κοινωνία των πολιτών ε, κολλείεται η κυρία Κρέτσου και μας ζήτησε να αναβάλω αυτό το σημείο. Οπότε, αν δεν έχετε αντίρρηση, συζήτηση για το θέμα αυτό αναβάλλεται για τις 16 ε, Σεπτεμβρίου. Αλλά δεν τροποποιείται το χρονοδιάγραμμα της έκθεσης Κρέτσου. Θα ψηφίσουμε δηλαδή στις 17 Σεπτεμβρίου, ενώ η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών λήγει στις 29 Ιουλίου το μεσημέρι. Ο κύριος Δέβα ε, δυστυχώς ε, δεν μπόρεσε να έρθει τελευταία στιγμή του συνέβη οπότε θα πρέπει να αναβάλουμε και την ε, δική του γνωμοδότηση για τις πληροφορίες που αφορούν τη μεταφορά ε, χρημάτων στην επόμενη συνεδρία που θα γίνει 16 και 17 Σεπτεμβρίου. Βέβαια, η 4η Σεπτεμβρίου στις 6 το βράδυ θα παραμείνει ως προθεσμία για την κατάθεση των απολογιών. Μία διόρθωση και για το σημείο 14 που προβλέπεται στην ημέρησια διάταξη θα συζητήσουμε ε, για, την, για τη διάσκεψη του κλίματος της Βαρσοβίας του Νοεμβρίου και κυρίως πώς θα συμβάλλουμε στην ε, κατάρτιση του ψηφίσματος ε, για την διάσκεψη αυτή για το κλίμα που θα γίνει στη Βαρσοβία. Άλλα σχόλια υπάρχουν και παρατηρήσεις για την ημέρηση διάταξη. Αν δεν υπάρχουν, εγκρίνεται η ούτως η μέρη σε διάταξη και περνούμε στην έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης μας συνεδρίασης, δηλαδή της 8 η και 9 η Ιουλίου του 2013. Αν έχετε παρατηρήσει για τα πρακτικά, θα, θα πρέπει να τις διαβιβάσετε στη γραμματεία πριν το τέλος της συνεδρίασής μας. Είδε μη, τα πρακτικά θα θεωρηθούν ως συγκεκριμένα. Σημείο 3. Ανακοινώσει της Προέδρου δεν υπάρχουν. Έχετε λάβει τις συστάσεις και τις αποφάσεις ε, της συνεδρίας των συντονιστών της 9ης Ιούλιου του 2013. Αν έχετε παρατηρήσεις για την έκβαση της συνεδρίας των συντονιστών, παρακαλώ να τις ε, κοινοποιήσετε στη γραμματεία πριν το πέρας της συνεδρίασης. Οι ΔΕΜΗ ε, θα εγκριθούν οι συστάσεις και αποφάσεις των συντονιστών αμετάβλητες. Ανακοινώσει επιτροπή δεν υπάρχουν. Για την ώρα των ερωτήσεων δεν έχουμε λάβει καμία ερώτηση, οπότε περνάμε στι εκθέσει επί τη ουσία. Το σημείο 7 πρώτα ε, που αφορά τις γυναίκες με αναπηρία. Η συντάκτρια της γνωμοδότησης είναι η κυρία Κρέτσου, αλλά όπως σας είπε κολλείεται για σήμερα και δεν θα μπορέσει να μας υποβάλει την έκθεσή της. Την αντικαθιστά ο κύριος Μαρτίνης, τον οποίο και δίνω μέσα το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αισθάνομαι ιδιαίτερα ευτυχής για την ευκαιρία που μου δίνεται να κηρύξω εγώ το εναρκτήριο λάκτισμα με το πρώτο θέμα επί της ουσίας αυτής της νέας φάσης των δραστηριοτήτων της Επιτροπής μας και να σας επιβεβαιώσω ότι όντως η κυρία Κρέτσου, που είναι η συντάκτρια της γνωμοδότησης για το θέμα γυναίκες με αναπηρία, δεν μπόρεσε να παραστεί. Ε, μάλιστα ζητά συγγνώμη για την απουσία της και μου ζήτησε να σας παρουσιάσω τις παρατηρήσεις της για τη γνωμοδότηση και μάλιστα θα διαβάσω τις ε, σημειώσεις της στα αγγλικά γιατί σε αυτή τη γλώσσα τις έχω λάβει. Γι' αυτό και θα μιλήσω στα αγγλικά όπως έκανε και η κυρία Κρέτσου για να μην την προδώσω στην ε, παρουσίαση των απόψεών της. Ξεκινάει λοιπόν η κυρία Κρέτσου λέγοντας ότι το θέμα αυτό είναι πολύ ευαίσθητο, μεταξύ άλλων γιατί αφορά τη ζωή πάνω από ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων. 80% αυτού του δισεκατομμυρίου ανθρώπων απαρτίζεται από ανθρώπους που ζουν σε αναπτυσσόμενες χώρες. Έτσι η πρόσβασή τους ε, στην υπηρεσίε στις υπηρεσίες υγείας ε, είναι δύσκολη και μάλιστα υπάρχει πρόβλημα και στην πρόσβαση στην εκπαίδευση. Οπότε ε, οι άνθρωποι αυτοί αντιμετωπίζουν και οικονομικές δυσκολίες και δύσκολα εντάσσονται στην αγορά εργασίας. Αντιμετωπίζουν και πολλές προκλήσεις ό,τι αφορά την πρόσβασή τους στην απονομή της δικαιοσύνης ή της δικαστικής αρρωγής, η νομικής αρρωγής σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων τους. Οπότε, γυναίκες που έχουν αναπηρίες ε, αντιμετωπίζουν πολύ περισσότερα προβλήματα από τις υπόλοιπες γυναίκες και μάλιστα παντού στον κόσμο. Το πρόβλημα αυτό όμως γίνεται πιο οξύ στις αναπτυσσόμενες χώρες. Εκεί πραγματικά είναι τραγική κατάσταση των γυναικών με αναπηρία. Και εμείς ε, ενδιαφερόμαστε κυρίως για την κατάσταση σε αυτές τις χώρες, αναπτυσσόμενες. Είμαστε Επιτροπή ανάπτυξη άλλωστε. Πολλές είναι οι ενισότητες, λοιπόν ε, που πλήττουν ε, τις γυναίκες με αναπηρία και έχουν μεταφράζονται σε πολλά μειονεκτήματα και δυσμενή μεταχείριση ό,τι αφορά την πρόσβαση στη στέγαση, στην επαγγελματική κατάρτιση, στην δανειοληψία ή στους παραγωγικούς πόρους. Και μάλιστα η τροτότητα αυτών των γυναικών ε, είναι ακόμη πιο μεγάλη γιατί είναι πολύ πιο εκτεθειμένες ε, σε σεξουαλική παρενόχληση, εκμετάλλευση και η δυσμενής πρόσβαση του στη δικαιοσύνη οξύνει ακόμη περισσότερο το φαινόμενο αυτό. Γι' αυτό και η συγγήτριά μας, η Κορίνα Κρέτσου, ε, υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να δώσουμε περισσότερα δικαιώματα στις γυναίκες με αναπηρία, να τις ενημερώσουμε καλύτερα και να άρουμε τα εμπόδια προκειμένου να διάγουν και αυτές ένα φυσιολογικό βίο θέλουμε μία προσέγγιση ε, που θα λαμβάνει υπόψη στην ισότητα των φύλων και τα προβλήματα των ανθρώπων με αναπηρία και ε, να περιλάβουμε τα προγράμματα μείωσης της φτώχειας, τα γεωγραφικά προγράμματα που έχουμε, καλύπτοντας ιδιαίτερα τις γυναίκες με αναπηρία. Η κυρία Κρέτσου τονίζει επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να στηρίξει τις προσπάθειες των ε, εταίρων σε ό,τι αφορά την κατάρτιση κατευθυντηρίων γραμμών για την απασχόληση, ώστε να περιλαμβάνονται τα θέματα ισότητας και στην ε, κυριότητα της ε, γης και να το και οι γυναίκες με αναπηρία στα θέματα αυτά. Η Κορίνα θεωρεί ότι θα πρέπει να δώσουμε πιο αποτελεσματική μάχη κατά της διακριτικής μεταχείρισης που υπόκεινται οι γυναίκες αυτές με πιο ευρεία πρόσβαση στην πρόσβαση και συμμετοχή των οργανώσεων ε, των ανθρώπων με αναπηρία στις εθνικές και διεθνείς ε, διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Η κυρία Κρέτσου ευχαριστεί και τη Γραμματεία για τη βοήθειά της και όλους μας για την κατανόηση, τους, για την κατανόηση που δείχνουμε σε ό,τι αφορά τη ζήτηση αυτού του σημείου ερήμη της, ε, τη απουσία της. Περιμένει πάντως διακάως τις τροπολογίες σας μέχρι αύριο το μεσημέρι από ό,τι ξέρω που και η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ όλους για την προσοχή που δείξατε για το θέμα αυτό. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ. Αυτά εκ μέρους της συγκήτριας της κυρίας Κρέτσου. Ευχαριστούμε κύριε Μαρτίνες. Η ε, κυρία Κρέσ. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ εξαιρετική δουλειά έκανε η συνάδελφος, βεβαίω και δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε ότι υπάρχουν ανισότητες και ακόμη χειρότερα γίνεται τα πράγματα και στην Ευρώπη και αλλού για τις γυναίκες με ειδικές ανάγκες και ακόμη περισσότερο στι αναπτυσσόμενε χώρες. Ακριβώς πρόκειται για κάτι το οποίο κορυφώνεται ε, οι γυναίκες αυτές οι οποίες υφίστανται τις ε, ανισότητες, οι ανάπηρες γυναίκες ακόμα χειρότερο και στις αναπτυσσόμενες χώρες ακόμα χειρότερα είναι τα πράγματα έχουν ακόμα ένα εμπόδιο να ξεπεράσουν δηλαδή οι γυναίκες αυτές οπότε και δεν μπορεί η πολιτική μας ομάδα παρά να συμφωνήσει ότι θα πρέπει αυτό το σημαντικό θέμα να αποτελεί βασικό στόχο ε, αναπτυξιακό για τη χιλιετία και να αποτελέσει άξονα στην πολιτική ανάπτυξη, ιστής πολιτικής ανάπτυξη και βέβαια ε, να δούμε τι θα πει η υπηρεσία εξωτερική δράση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσον αφορά το θα πρέπει να υπάρχει κάποιο είδου εποπτεία, κάποιο είδου έλεγχο, κάποιο είδου αξιολόγηση αυτών των πολιτικών για να διαπιστώσουμε εάν είναι αποτελεσματικές και όπως και για άλλα ζητήματα και εν προκειμένου θεωρούμε ότι θα πρέπει να χαρακτηριστεί το θέμα αυτό εγκάρσιο και να έχουμε μια προσέγγιση συνεπή. Άρα θα πρέπει η Ευρώπη να βοηθήσει κάτι να κάνει και να αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες ευρωπαϊκές αλλά και σε εθνές επίπεδο για τα θέματα των δύο φίλων και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 θα δώσω τη σκητάλη στον συνάδελφο από την ΤΕΦΚΟ, αλλά πάντως εμεί από πλευρά τη υπηρεσία δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε αυτή την πρωτοβουλία. Και με τα όσα έχουν αναφερθεί, με τα όσα έχουν προταθεί και με τις τροπολογίες, να σε εξηγήσω γιατί. Έχουμε προσυπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή την διεθνή συνθήκη και έχουμε αναλάβει και εμεί υποχρεώσει, οι οποίες συγκεκριμένα αφορούν το πώς θα ε, βοηθήσουμε τους ε, αναπήρους στα πλαίσια πολιτικού διαλόγου και διαλόγου για τα ανθρωπινά δικαιώματα. Οπότε και θα πρέπει προοδευτικά ε, για σιγά σιγά να έρθουμε σε επαφή με τους φορείς αυτούς όσον αφορά τα διάφορα φύλλα, τους αναπήρους και ήδη έχουμε εξετάσει κάποια σχετικά προγράμματα να αναπήρους να συνεχιστεί σε ένας ανοιχτός διάλογος με τις αρχές. Να πιέσουμε τις αρχές και τις κυβερνήσεις να προσυπογράψουν αυτή τη διεθνή συνθήκη για το σεβασμό των δικαιωμάτων των αναπήρων. Θα πρέπει όλες οι κυβερνήσεις επομένως να βοηθήσουν στην υλοποίηση αυτής της ε, συνθήκης. Και εδώ τώρα μιλούμε πιο συγκεκριμένα για τις ανάπηρες γυναίκες, οπότε και θα πρέπει να τονιστεί και αυτό. Άρα, συμφωνούμε με όλες τις προτάσεις που διατυπώθηκαν. Και θα συνεχίσουμε να θέτουμε το ζήτημα στα πλαίσια του συνεχούς διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε επίσης στο χάρτη των δικαιωμάτων το άρθρο 8, οπότε και όποτε υπάρχει θέμα ανθρώπινου δικαιώματος θα τονίζεται το τι γίνεται με τις, ε, με τις ε, ανάπηρες γυναίκες. Και τώρα δίνουμε την ε, σκητάλη στον κύριο Τάιλερ από την ΤΕΦΚΟ. Ευχαριστώ πολύ. Όπως υπόθηκε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας από τους μεγαλύτερους ε, ευεργέτες και προσπιστές του Συμφωνού για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία, φροντίζοντας για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων για τους ανθρώπους με αναπηρία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευθεί να συμπεριλάβει λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους και λαμβάνουμε τα κατάλληλα βήματα έτσι ώστε σταδιακά να πραγματοποιηθούν οι δεσμεύσεις μας. Ωστόσο, θα μπορέσουμε να λάβουμε καλύτερα υπόψη και να υλοποιήσουμε τις προδιαγραφές αυτές εάν υπάρξει και η κατάλληλη ανταπόκριση. Για παράδειγμα, η αναπηρία έχει συμπεριληφθεί ως ένα εγκάρσιο ζήτημα στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ψηφίστηκε από την Επιτροπή το Σεπτέμβριο του 2011 και στις ε, νέες κατευθυντήριες ε, γραμμές για τον προγραμματισμό. Έπειτα, έχουμε συμπεριλάβει τις, ε, τους ανθρώπους με αναπηρία στις κατευθυντήριες γραμμές της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, φροντίζουμε να συλλέγουμε στοιχεία αναχώρα για τους ανθρώπους με αναπηρία και να συμπεριλαμβάνουμε τα στοιχεία αυτά σε αξιολογήσεις να προωθούμε την ενεργό συμμετοχή των ανθρώπων με αναπηρία σε οργανισμούς. Διασφαλίζουμε την πρόσβαση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις υπηρεσίες σε σχετικές για τους ανθρώπους με αναπηρία και στην ευαισθητοποίηση και ενίσχυση της επικοινωνίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει ένα πρόγραμμα κατάρτιση σε συνεργασία με την Υπηρεσία Εξωτερική Δράση για ενισχυμένη συνεργασία. Το 2012, το Νοέμβρη, άρχισε το πρώτο στάδιο του προγράμματο που στόχο έχει να ενισχύσει, όπω είπαμε, την ε, ενημέρωση και την συνεργασία. Και στο διαδίκτυο επίσης. Τώρα, όσον αφορά το σημείο 5 για την ε, στήριξη που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις ε, χώρες εταίρους για την εφαρμογή της, ε, της, των διατάξεων στην εθνική τους νομοθεσία. Να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει ένα νέο πρόγραμμα, το CERCER, το οποίο θα παρέχει εμπειρογνωμοσύνη σε όλες τις χώρες εταίρους για την ανάπτυξη συστημάτων κοινωνικής προστασίας. Αυτό είναι κάτι αναγκαίο και θα βοηθήσει στην ε, σύνταξη κατάλληλη νομοθεσία, Ταυτόχρονα, όσον αφορά τη στήριξη ανθρώπων με αναπηρία, ιδιαίτερα των γυναικών με αναπηρία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα Τέξει ένα πρόγραμμα φέτος που θα δώσει προσοχή και βάρος στην πρόσβαση των ε, μειονεκτούντων ανθρώπων στις ε, υπηρεσίε. Το πρόγραμμα αυτό πρέπει να συνάδει με την ε, διατάξει του Συμφώνου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το, ιδιαίτερα το άρθρο 28 για τα στάνταρ ζωή. Τώρα, όσον αφορά την ιδιοκτησία, υπάρχουν πολλά προγράμματα που επικεντρώνονται στην Αφρική και στόχο έχουν την καταπολέμηση του γυναικείου αναλφαβητισμού και την προώθηση της ιδιοκτησίας γης από γυναίκες με αναπηρία και στόχος ε, είναι η μείωση των ανισοτήτων στην περιοχή αυτή. Επίσης, η αναπηρία αντιμετωπίζεται ως ε, θέμα εγκάρσιο και αναφέρεται σε όλες τις προτάσεις που έχουμε για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μαρτίνες, έχετε το λόγο, αν θέλετε, για να ολοκληρώσουμε. Αν το επιθυμείτε φυσικά. Όχι, απλώς ήθελα να πω ότι Πιστεύω ακράδαντα ότι θα είναι αποτελεσματική αυτή η γνωμοδότηση και η έκθεση και χαίρομαι ότι και η συγκεκριμένη επί της ουσίας, ε, η κυρία Βέρμαν, είναι πολύ σοβαρή, σοβαρός άνθρωπος ε, που ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το θέμα αυτό, γι' αυτό και με βέβαιος ότι το έργο θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Σίγουρα θα συμπληρώσουμε την κύρια έκθεση με τη δική μας γνωμοδότηση, με τη γνωμοδότηση δηλαδή της κυρίας Κρέτσου. γιατί και εμείς έχουμε να πούμε πολλά για το πρόβλημα των γυναικών με αναπηρία στις αναπτυσσόμενες χώρες. Πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Και τα σχόλια της Επιτροπής και της ΕΙΕΔ με χαροποίησαν. Γιατί πραγματικά πιστεύω ότι υπάρχει δυνατότητα για συνεργασία και πρόοδο. Και συμφωνώ απόλυτα και με την κυρία Γκρέσ. Γιατί έχουμε αυτή την επαρλία γεγονότων και άνθρωποι που ούτως ή άλλως ε, υφίστανται δυσμενή διαχείριση και σε φυσιολογικές συνθήκες, ε, στην περίπτωση αυτή είναι σε ακόμη χειρότερη θέση στις αναπτυσσόμενες χώρες και στις γυναίκες που έχουν μια, κάποια αναπηρία. Είναι σημαντικό λοιπόν να εγκύπτουμε στο πρόβλημα αυτό και να ασκήσουμε και πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να σημειώσει πρόοδο. Είναι ενδιαφέρον λοιπόν και πολύ σημαντικό που ασχολούμαστε με το θέμα αυτό. Και πολύ ελπιδοφόρο άλλωστε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να σας υπενθυμίσω, όπως είπε ο κύριος Μαρτίνες, ότι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών λίγη αύριο στις 12 το μεσημέρι. Η ψηφοφορία θα γίνει στις 17 Σεπτεμβρίου. Και περνάμε στο σημείο 8 της ημέρης της διάταξης. Την παρουσίαση της γραμμοδότησης τη ε, έκθεση της Επιτροπή Υπολογισμών ό,τι φορά τη χορήγηση εγγύηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν επενδυτικά έργα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για νομοθετική γνωμοδότηση. Συντάκτης της είναι ο κύριος Πρέντα. Ε, δυστυχώς ο κύριος Πρέντα δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα γιατί είναι επικεφαλής αντιπροσωπείας παρατηρητών για τις εκλογές ε, στη Γουινέα Κόνακρη και έπρεπε να μεταβεί εκεί. Γι' αυτό θα δώσω το λόγο στην κυρία Μισελ Στίφλερ για να μας παρουσιάσει το σχέδιο γνωμοδότηση στη θέση του κυρίου Πρέντα. Κύριος Πρέντα, ζητά συγγνώμη που δεν μπόρεσε να παραστεί ούτως ώστε να παρουσιάσει το σχέδιο έκθεσης οπότε και εγώ απλώς θα σας διαβάσω το κείμενο του γιατί είναι το πιο μεγάλο ε, ίδρυμα τραπεζικό που μπορεί να παράσχει αυτές τις εγγύησεις τόσο ώστε να υποστηρίξει τις δραστηριότητες μας στις τρίτες χώρες. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η υπόθεση για την Επιτροπή μας, διότι έτσι θα μπορούσαμε να δούμε πώς η ΕΤΕ πρόκειται να λειτουργήσει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επόμενη επταετία. Και έχουμε επομένως αυτό το νομοθετικό πλαίσιο για τις δραστηριότητες της ΕΤΕ στις τρίτες χώρες. Αυτό βελτιώθηκε σύν χρόνο και σημαντικά συνέβαλε σε αυτό το κοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι είναι θετικές αυτές οι εξελίξεις και πρόκειται για αυτή την εντολή όσον αφορά τη χρηματοδότηση, όσον αφορά την άσκηση της εξωτερικής οργής όπως ορίζεται στο αρθρικό της συνθήκης και επίσης έτσι θα εξασφαλιστεί η συμμετοχή του κοινού. Άλλα στοιχεία που πρέπει να αναφέρουμε είναι τι θα κάνει η ΕΤΕ για τους λιγότερο φερέγγιους δικαιούχους. Όπως επίσης και το πλαίσιο που ορίστηκε για την δημοκρατία και έτσι η ΕΤΕ θα είναι πιο αποτελεσματική για να βοηθήσει την αναπτυξιακή πολιτική μας. Για την Επιτροπή μας είναι πάρα πολύ σημαντικό οι ενέργειες της ΕΤΕ στα πλαίσια της εξωτερικής εντολής θα πρέπει να υποστήξουν αυτούς που έχουν περισσότερο ανάγκη και να υπάρχει ένας αντίκτυπος για την ανάπτυξη. Πολύ σημαντικό επομένως να εξασφαλίσουμε την προσαρμογή αυτής της ε, πολιτικής με τις πρόσφατες εξελίξεις. Ε, επίσης να δούμε πώς θα χτενίσουμε, πώς θα βελτιώσουμε τις διατάξεις για τις ε, ΜΜΕ και έτσι να υπάρχει αντίκτυπο στην ανάπτυξη και διαφάνεια. Επίσης λέει ο Ισηρής ότι θα πρέπει αυτή η εντολή να να πώς ανθρώπινα δικαιώματα και να έχει επιπτώσεις και σε τοπικό επίπεδο, οπότε να υπάρχει ένας εποπτικός μηχανισμός για να λέγεται εάν όλα αυτά είναι σύμφωνα με το άρθρο 21 και επίσης τονίζει ο Ισπηδής ότι για να συντάξει αυτή την έκθεση πιέστηκε πάρα πολύ από πλευράς χρόνου και άρα έτσι θα πρέπει να υπάρξουν διορθωτικές κινήσεις μέσω των ε, τροπολογιών και άρα περιμένει τη βοήθεια των συναδέλφων. Πρόεδρος, ευχαριστούμε και τώρα το λόγο κυρία Pardon. Με ακούτε τώρα. Ωραία. Η αρχική πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι αρκετά καλή. Ο συγητής μάλιστα τη βελτίωσε και διευκρίνησε αυτά τα τρία θέματα, μείωση της φτώχειας, δημοκρατία και κατάσταση στον ιδιωτικό τομέα. Είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι λοιπόν με την γνωμοδότηση. Θα ήθελα να υπενθυμίσω μερικές βασικές αρχές που θα πρέπει να τονιστούν. Η πρώτη αφορά την ανάγκη ευθυγράμμιση με τις αναπτυξιακές πολιτικές που προωθούνται από τις ίδιες αναπτυσσόμενες χώρες. Θα πρέπει δηλαδή να σεβαστούμε εδώ την κυριαρχία των αναπτυσσόμενων χωρών σε ό,τι φορά τη χάραξη αυτών των αναπτυξιακών πολιτικών. Δεύτερο σημαντικό θέμα τα κριτήρια επιλογής ε, και τα, στα σχέδια και η αξιολόγησή τους θα πρέπει ε, να προσανατολίζονται στο τελικό αποτέλεσμά τους ό,τι φορά την ανάπτυξη. Και φυσικά θα πρέπει να ευνοήσουμε τις τοπικές επιχειρήσεις. Αυτό είναι σημαντικό αν θέλουμε αυτά αποτελέσματα σε θέματα ανάπτυξης. Επίσης, μας ενδιαφέρει και η διαφάνεια των χρηματοοικονομικών στοιχείων, των χρηματοπιστωτικών στοιχείων που χορηγούν οι επιχειρήσεις, προκειμένου να καταπολεμηθεί το φαινόμενο της φοροδιαφυγής. Θα υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες, κυρίως ό,τι αφορά τα χρηματοοικονομικά θέματα και τους ε, μεσάζοντες, τη φοροδιαφυγή ή τα μέτρα καταπολέμησης της διαφθορά της απάτης. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μπέργμαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας α, ξαναβλέπω με ιδιαίτερη χαρά μετά τις α, θερινές διακοπές που συνήθως είναι πολύ σύντομες. Έχω κάποιες α, παρατηρήσεις εκ του κυρίου Λάστρα που είναι ο σκιώδης ηγητής για το θέμα αυτό. Η ΕΤΑ είναι ένα από τα πιο σημαντικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα παραμείνει σημαντική λόγω της ε, συνεισφοράς στην ανάπτυξη, η οποία δεν γίνεται χωρίς την χρηματοπιστωτική δραστηριότητα. Καλωσορίζουμε λοιπόν τη γνωμοδότηση τη έκθεση για τον προπολογισμό, ιδιαίτερα όσον αφορά τη χορήγηση εγγυήσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την κάλυψη ζημίων. Αυτό εξάλλου είναι κάτι το οποίο συζητούμε από το 2010 ε, αν και η πρόταση αυτή δεν συμπεριλαμβάνει όλε τι τροποποιήσει που πρότεινε το Κοινοβούλιο και ενέκρινε με την πρώτη ανάγνωση στην ολομέλειά του μετά τι διαπραγματεύσει, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατάφερε ε, να, να ληφθεί σοβαρά υπόψη η ε, πρότασή του, ιδιαίτερα όσον αφορά την διαφάνεια, την αναφορά, τα ανώτατα όρια, την ευελιξία, την συνεισφορά στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την μείωση της φτώχειας και την ερεσιμότητα μεταξύ άλλων. Καλωσορίζουμε λοιπόν την πρόταση του εισηγητή που προτρέπει την ε, την εστίαση στις ε, χώρες που έχουν περισσότερη ανάγκη. Και ιδιαίτερα όσον αφορά την αύξηση της ε, διαφάνειας και της λογοδοσίας. Ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ τον εισηγητή. Σας ευχαριστώ κύριε Γκέρενς. Ευχαριστώ. Εγώ έχω κάποιες ερωτήσεις τεχνικού χαρακτήρα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η γνωμοδότηση αυτή ενθαρρύνει την ΕΤΕΠ να δανείσει χρήματα σε λιγότερο φερέγγιους αποδέκτες. Σε ό,τι αφορά αυτή την λυπή φερεγγιότητα, ποια είναι τα εφαρμοστέα κριτήρια Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής. Και οι χώρες που δικαιούνται την δημοσιονομική υποστήριξη θεωρούνται φερέγγιες, ενώ αυτές που δεν δικαιούνται δημοσιονομική συνδρομή ε, δεν θεωρούνται φερέγγιες. Μια διευκρίνηση θα ήθελα προς το θέμα αυτό. Δεύτερη ερώτηση. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπορεί να δανείζει σε χώρες, ε, σε θεσμικά όργανα, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. Και αυτή η μειωμένη φερεγκαιότητα που αναφέρει η έκθεση αφορά και τον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα τύχει ε, της ε, χορήγης εγγύησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να αντιμετωπίσουν κινδύνους για δάνειο που χορήγησε σε, στον ιδιωτικό τομέα. Τρίτο. Ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σε περίπτωση ε, δανείων σε χώρες ε, στις οποίες δραστηριοποιείται και παρέχει συνδρομή, γιατί στις χώρες αυτές ε, έχουμε και τοπικές αναπτυξιακές τράπεζες, όπως την Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα επενδύσεων δίνει προτεραιότητα στις τοπικές τράπεζες, στην Αφρικανική Αναπτυξιακή Τράπεζα για παράδειγμα ή στην Διαμερικανική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Γιατί υπάρχουν και τέτοιοι μηχανισμοί με πολύ σημαντικά κονδύλια πολύ συχνά. Οπότε ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Γιατί είναι ιδιαίτερα συνετή συνήθως και τετοιοι μηχανισμοι με πολυ σημαντικα κονδυλια πολυ συχνα οποτε ποια ειναι η θεση της ευρωπαικης τραπεζας επενδυσεων γιατι ειναι ιδιαιτερα συνετη συνηθω και ενδιαφερεται να κρατήσει το τριπλό της α από του οίκου αξιολόγηση, οπότε ποια θα είναι η θέση σε τέτοια περίπτωση. Αυτές είναι οι ερωτήσει. μου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να θέσω μια ερώτηση στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Γιατί είχαμε πάει με την Καθρίν Γκρέ και την κυρία Λούνατσεκ στη Βραζιλία, στο κρατήδιο Παρά, ε, επισκεφθήκαμε το φράγμα του Μπελομόντα και την ολέθρια, τις ολέθριες ε, επιδράσεις που έχει στο περιβάλλον. Αλλά όχι μόνο στο περιβάλλον και στους τοπικούς πληθυσμούς. Το σχέδιο ε, ε, κατασκευής αυτού του φράγματος, που είναι το τρίτο μεγαλύτερο φράγμα του κόσμου, ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα δηλαδή, χρηματοδοτείται από την Βραζιλιάνικη Τράπεζα Ανάπτυξης. Και έμαθα ότι και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων από ό,τι ξέρω δάνεισε 500 εκατομμύρια σε αυτή την ε, Βραζιλιάνικη Τράπεζα Ανάπτυξης. Ερωτώ λοιπόν, υπήρξαν κάποιες ασφαλιστικές δικλίδες ώστε ε, σε καμία περίπτωση κοινοτικά κονδύλια να μην ε, αξιοποιηθούν για την κατασκευή αυτού του φράγματος που δεν θα εξυπηρετήσει καμία περίπτωση τον τοπικό πληθυσμό, αλλά τις πολυεθνικές που θα ε, εκμεταλλευτούν τα γειτονικά ορυχεία. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της ΕΤΕΠ, στον κύριο Αλεξάνδρο Καράνοφ. Ε, Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις και τις απόψεις σας και ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία που μας δώσατε να παρευρεθούμε και να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας. Ε, γενικά καλωσορίζουμε την συμμετοχή του Κοινοβουλίου για την εξωτερική αυτή έντολη. Πρόσφατα είχαμε και την ενδιάμεση αναθεώρηση της εφιστάμενης εξωτερικής εντολής και αυτή εδώ η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο μας βοήθησαν πάρα πολύ με τις προτάσεις τους που ενσωματώθηκαν στις δραστηριότητές μας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Όπως ίσως γνωρίζετε, αυτό σημαίνει περισσότερη προσοχή στις επιπτώσεις των ε, δραστηριοτήτων μας, ιδιαίτερα από πέρυσι. Έχουμε το πλαίσιο μέτρησης αποτελεσμάτων, ε, έχει τεθεί σε εφαρμογή και με αυτό μπορούμε να αξιολογήσουμε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων μας ε, και ποιες είναι οι επιπτώσεις που αναμένονται όσον αφορά την ανάπτυξη λοιπόν αυτών των δραστηριοτήτων και όλες τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις σε όλους τους ε, τομείς. Όπως ε, αναφέρατε, για τις ανάγκες, πιστεύω και εγώ πως οι ανάγκες ε, των χωρών αυτών είναι τεράστιες, ιδιαίτερα όσον αφορά τις επενδύσεις που είναι αναγκαίες στον ιδιωτικό τομέα, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε έργα υποδομής αλλά και σε άλλους τομείς, όπως για παράδειγμα την υγεία και την παιδεία. Υπάρχουν περίπου 70 χώρες που καλύπτονται από αυτήν την εντολή. Για το λόγο αυτόν, λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνουμε ενδείξεις και πληροφορίες από όσους χαράσουν πολιτική και ταυτόχρονα να μπορούμε να εφαρμόσουμε και όλες τις απαιτήσει και να πληρούμε τις ε, προϋποθέσεις, διότι μιλάμε για δάνεια, για επενδύσεις, για δανεισμό γενικότερα. Τώρα, όσον αφορά τις ε, προτεραιότητες ε, της πολιτικής, μπορούν να παρέχονται και από το Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, όσον αφορά τα ανώτατα όρια. Πιστεύουμε πως εξαιτία των περικοπών που έχουν γίνει έχει παρατηρηθεί μία μείωση στην στο εύρος της εντολής, το ποσό που μπορούμε να δανείσουμε. Μπορούμε να, δανείσουμε περίπου, να διαθέσουμε περίπου 30 δισεκατομμύρια, σκοπεύουμε να τα χρησιμοποιήσουμε, αλλά για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο το ποσό αυτό θα μειωθεί στα 25 δισεκατομμύρια. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι ανάγκες είναι τεράστιες, Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα όσον αφορά τι χώρε γειτονία αλλά και τι ε, χώρε που βρίσκονται σε πρωταξιακό στάδιο, έχει μεγάλο σημαντικό ρόλο να παίξει. Ταυτόχρονα όμω γνωρίζουμε το πόσο μικρό είναι το περιθώριο για ευελιξία που έχουμε. Γι' αυτό λοιπόν εάν μπορούμε να ανακατανείμουμε κάποια κονδύλια, έστω και 100 εκατομμύρια, θα μπορέσουμε να τα αξιοποιήσουμε με το βέλτιστο τρόπο. Θα μπορούσαμε λοιπόν να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να επεξεργαστούμε αυτό το σημείο έτσι ώστε να μεγιστοποιήσουμε τις δυνατότητες δανεισμού μας. Ιδιαίτερα, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για να δημιουργεί προστιθέμενη αξία την οποία θέλουμε. Τώρα, υπήρξαν αναφορές στη δημοκρατία και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Φυσικά και αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά σημεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι πάρα πολύ σημαντικό να λαμβάνουμε ενδείξεις από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και πληροφορίες και να τις ερμηνεύουμε. Αυτές να τις συμπεριλαμβάνουμε στην αξιολόγηση των χωρών που μπορούν να λάβουν αυτήν την βοήθεια έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να μπορεί να δραστηριοποιηθεί σε αυτές τις χώρες. Και αν μια χώρα δεν θεωρείται κατάλληλη για να λάβει ευρωπαϊκή βοήθεια πλέον, μπορεί αυτή να αφαιρεθεί από τον κατάλογο μέχρι να γίνει αξιολόγηση όσον αφορά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Αυτό που εμείς κάνουμε είναι στηριζόμαστε στο πλαίσιο αυτό για τις ε, λειτουργίες μας και στηριζόμαστε και στην ε, βοήθεια από τα άλλα θεσμικά όργανα για να το πράξουμε αυτό. Θα γίνει λοιπόν αξιολόγηση αντικτύπου βάση της οποίας θα κρίνουμε εάν ένα project μπορεί να συνεχιστεί. Παρομοίως και με, τα, και με τις επιπτώσεις περιβαλλοντικού αντικτύπου. Πρέπει λοιπόν να ξέρουμε τι περιμένουμε και με τι έχουμε να κάνουμε. Έχουμε πολύ μικρό αριθμό προσωπικού σε σχέση με τις ε, άλλες ε, τράπεζες περιφερειακής ανάπτυξης που ανέφερε ο κύριος Εκόρενς και έχουμε το 1 δέκατο των κονδυλίων για να βελτιστοποιήσουμε την, ε, τις επιπτώσεις των δανείων μας. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε, διότι αυξάνονται οι απαιτήσει για εμάς και φυσικά αυτό είναι καλοδεχούμενο, αλλά από την άλλη είναι σημαντικό να καταλάβουμε και τι αυτό συνεπάγεται. Η πρόταση αυτή παρέχει εγγύηση για κάλυψη του κινδύνου. Αυτά στον δημόσιο τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα όμως υπάρχει κάλυψη, αλλά μόνο σε περίπτωση χρεοκοπίας από πολιτικούς ε, παράγοντες και όχι από άλλους παράγοντες. Εκεί δεν καλύπτουμε τις περιπτώσεις αυτές. Μόνο σε περίπτωση, για παράδειγμα, εμφυλίου πολέμου, πολιτικών ε, αναταραχών παραβίαση συνθήκων κτλ. Αυτά υπάρχουν στις ε, λεπτομέρειες στο έγγραφο των εγγύσεων που προβλέπονται από την ΕΤΕ. Τώρα, όσον αφορά την ε, περισσότερο άμεση επίδραση στην ανάπτυξη, αυτό θα αυξηθεί αν αλλάξει το επιχειρηματικό μοντέλο, αν αλλάξει η χωρητικότητα, αν αλλάξουν οι δυνατότητες απορρόφησης ε, των κονδυλίων. Γι' αυτό το θέμα είμαστε ανοιχτοί προς συζήτηση. Τέλος, Είμαστε επίσης ανοιχτοί σε προτάσεις για βελτίωση των ε, μέσων που διαθέτουμε. Έχει, έχουν βελτιωθεί πολλά συστατικά στοιχεία των ε, επιχειρησεών μας. Ε, ήδη ζητούμε πλήρη και απόλυτη διαφάνεια από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για δάνεια που λαμβάνουν από την ΕΤΕΠ. Και ήδη ζητούμε και από τις τράπεζες που έχουν το ρόλο μεσολαβητή να μας παρέχουν αυτές ε, τις ε, πληροφορίες. Ε, επίσης, αν θυμάμαι καλά και αν έχω το χρόνο, θα ήθελα να απαντήσω σε ορισμένες πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Λαμβάνοντα υπόψη το γεγονό ότι έχουμε χορηγήσει δάνεια σε λιγότερο φερέγγιες ε, χώρες, θα ήθελα να αναφερθώ στις χώρε που βρίσκονται στο παράρτημα. Να σας πω ότι εμείς εργαζόμαστε με βάση αυτές τις χώρε που αναγράφονται στο παράρτημα και αυτές ε, δανειοδοτούμε. Φυσικά, θα προσπαθήσουμε να εστιάσουμε τις επαρεμβάσεις μας στις χώρες στις οποίες μπορούμε να έχουμε τα μέγιστα δυνατά ωφέλη και αποτελέσματα. Και η Τράπεζα Επενδύσεων συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις χώρες αυτές ε, και για την ε, κατανομή των πόρων. Υπάρχει φυσικά μια σχέση ανάμεσα στην εφεργειότητα μιας χώρας και στο ποσό που διατίθεται από τον προϋπολογισμό για τη χώρα αυτή. Όσον αφορά την συνεργασία με άλλες ε, τράπεζες ανάπτυξης, να σας πω ότι μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποια, κάποιο ιδιαίτερο πρόγραμμα προτίμησης της ε, τράπεζας αυτές ή στην Ευρωπαϊκή Τραπέζα Επενδύσεων. Επίση, να σα πω ότι πολλά από τα project αυτά συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε συνεργασία με τι ε, περιφερειακέ τράπεζε ανάπτυξη. Έχουμε περισσότερο δηλαδή ρόλο παρατηρητή, αλλά δεν ζητούμε προτεραιότητα όσον αφορά τα έργα που χρησιμοποιούν κονδύλια μας. Επίσης έχουμε πολλές συμφωνίες ε, συνεργασίας, ε, συμφωνίες συγχρηματοδότησης με περιφερειακές ε, τράπεζες και όσον αφορά το ερώτημά σας για την Τράπεζα Ανάπτυξης της Βραζιλίας, όντως υπάρχει ένα ανοιχτό δάνειο 100 εκατομμυρίων, αλλά το δάνειο αυτό δεν έχει ακόμα απελευθερωθεί προς την τράπεζα αυτή της Βραζιλίας ε, λόγω ορισμένων ε, ζητημάτων που έχουν να κάνουν με τις ε, δημόσιες συμβάσεις. Διεξάγουμε εξονυχιστικούς ελέγχους, όμως θα επανέλθω με περισσότερες πληροφορίες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και τώρα κύριος Γκέρενς. Έχω μια συμπληρωματική πρακτική ερώτηση. Όταν ξεκινά αυτή η διαδικασία, δηλαδή να χορηγηθεί μια τέτοια εγγύηση. Ποιος έχει την πρωτοβουλία, η ΕΤΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και το πρώτο σενάριο είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνει ότι συμφέρει να χρηματοδοτήσει κάποιο πρόγραμμα, κάποιο έργο, μια που δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα, τότε λέτε στην ΕΤΕ να χορηγήσει ως δάνεια τα χρήματα που χρειάζονται ή μήπως η ΕΤΕ σαν δεύτερο σενάριο έχει τη δυνατότητα να πει έχουμε αυτό το έργο, το πρόγραμμα ενδιαφέρον είναι επιλέξιμο για κάποια εγγύηση την οποία θα χορηγήσει η Επιτροπή. Ισχύει το πρώτο, το δεύτερο σενάριο ή και τα δύο. Κύριε δικά να το λόγο. Αυτό γίνεται, ενεργοποιείται αιτήσει των εργολάβων των Σιπινόπουλων για τα περισσότερα μας δάνεια. Έτσι χορηγούνται. Μπορεί να ε, ασχολείται με αυτό κάποιο Υπουργείο, Υπουργείο Οικονομικών Ανάπτυξης κάποιας χώρας. Και συνήθως έτσι γίνεται πλευράς το Στον ιδιωτικό τομέα τώρα παρομοίως η εταιρεία η οποία θέλει να την δανείσει η ΕΤΕ. Οπότε υποβάλλει αίτηση ο εργολάβος εις δε τον ε, δημόσιο τομέα υπάρχει συνεχής διάλογος με τις ε, εν λόγω χώρες και την ΕΤΕ την εκεί αντιπροσωπεία οπότε κατά αυτόν τον διάλογο η χώρα διατυπώνει την ανάγκη την οποία έχει. Οπότε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει το κατά πόσον είναι ε, δέουσα η παρέμβαση της ΕΤΕ. Συνήθως πάντως είπαμε ο εργολάβος ε, ζητεί από την ΕΤΕ να του χορηγήσει το δάνειο και αυτό ισχύει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Και το λόγο έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Και στο παρελθόν έχουμε συζητήσει το πώς μπορούμε να συνδυάσουμε αυτά τα κεφάλαια από το EIF και από την ΕΤΕ. Βεβαίω προβλέπεται και αυτή η εγγύηση που αποτελεί τμήμα αυτής της χρηματοδότησης ούτω ώστε να διευκολύνουμε κάτι το οποίο θα ήταν τελείω δυνατό, δηλαδή το να μπορέσει η ΕΤΕ να στηρίξει ε, οικονομικά τα έργα, τα προγράμματα που χρειάζεται. Εδώ και δύο χρόνια ισχύει αυτό, όσον αφορά τη χρήση την αξιοποίηση αυτής της εγγύησης όπως ε, προελέχθη. Πολύ σημαντική υπόθεση. Είδε ότι που άλλαξε η αρχική πρόταση, δηλαδή να χρησιμοποιηθεί η εγγύηση όπου χρειάζεται. Αυτό τι σημαίνει. Ότι ενθαρρύνεται η ΕΤΕ να αναλαβεί το ρίσκο κάποιες χρηματοδότησης όπου χρειάζεται και Επίσης, θα πρέπει να συζητηθεί σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να αξιοποιηθεί η εγγύηση. Και ερχόμαστε τώρα σε αυτό το οποίο ρώτησε ο κ. Γκέρνς. Δεν είναι εύκολο να απαντηθεί η ερώτησή σας. Σε ποιες χώρες δηλαδή θα χρησιμοποιηθεί η εγγύηση και πώς θα συνδεθεί άμεσα με τις χώρες που έχουν δημοσιονομική υποστήριξη Επίση είναι το θέμα βιωσιμότητας του χρέους, σε κάποιες χώρες δηλαδή που δεν μπορούν να λειτουργήσουν αλλιώ. που δεν μπορούν να δανειστούν ή μπορούν να δανειστούν με υπερβολικά υψηλό επιτόκιο. Πάντω αυτό κρίνεται αναπερίπτωση. περίπτωση. Επίσης, σας τονίζω ότι συνεργαζόμαστε με την εταιρεία για τις εγγύσεις αλλά και για τις διάφορες άλλες διευκολύνσεις τα τελευταία χρόνια και σε αυτό το πλαίσιο γιατί καλύπτεται από τον προϋπολογισμό και από το Ταμείο Ανάπτυξης. Και επίσης, για να απαντήσω και κάποια άλλη ερώτηση, όσον αφορά αυτές τις διευκολύνσεις, εμπλέκονται διάφορα τραπεζοοικονομικά ιδρύματα όπως περιφερειακές τράπεζες. Και θεωρούμε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό πλεονέκτημα. Οπότε και ενθαρρύνουμε και την ε, ΕΤΕΝ αλλά και τις άλλες τράπεζες να εμπλακούν σε αυτή την προσπάθεια περισσότερο στο μέλλον. απαντήσαμε για τον ιδιωτικό τομέα, τώρα όσον αφορά την πρωτοβουλία για αυτά τα προγράμματα, αυτό συζητείται στα πλαίσια της πλατφόρμας Ένωσης για αυτό το, το μείγμα παρέμβασης. Και κατά το πρώτο εξάμεινο του ενεστώτος έτους είπαμε ότι θα ενθαρρύνουμε τις τράπεζες αλλά και την εταιρεία στο μέλλον. Ακόμη περισσότερο να εμπλέξουν τις αντιπροσωπείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την αρχή των κινήσεων αυτών. Αν δηλαδή υπάρχει κάποια τέτοια πρωτοβουλία από κάποιο εργολάβο, θα πρέπει αυτή εξ αρχή η αντιπροσωπεία της Ένωσης να ασχοληθεί και έτσι να υπάρξει στενή συνεργασία μεταξύ Κομισιών και ΕΤΕ για όλα τα έργα και προγράμματα. Όμως, η αντιπροσωπεία της ΕΕ προσεγγίζει την ΕΤΕ, εάν έχει κάποιο τοπικό γραφείο επιτόπου ή τόσο κατά κάποιο τρόπο, σύμφωνα με τις προτεραιότητες που έχουμε τάξει για, την, για τη χώρα την προκειμένα όσον αφορά την ανάπτυξη. Επίσης, κάποιος είπε κάτι για την φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. διάλογος σύντησε είναι συνεχής, δεν είναι εύκολο θέμα. Δεν είναι ξεκάθαρο το πλέγμα κανόνων που ισχύουν, ούτε τα όσα ισχύουν στα πλαίσια του όσα βοηθούν πάρα πολύ, άρα θα πρέπει να παρακολουθήσουμε την υπόθεση και την εξελιξή του αμέσως επόμενους μήνες. Και για τις ε, περιπτώσεις ε, επιχειρηματικών κεφαλαίων ή κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου τέλο πάντων, θα πρέπει να δούμε πώς θα αξιοποιήσουμε τους πόρους που υπάρχουν. Αυτά από πλευράς μου. Ο κύριος Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια. Εγώ είμαι συντάκτης γνωμοδότησης επί της οδηγίας για τη διαφάνεια ε, για τις, για τις μεγάλες επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Ο Μισελ Μπαρνιέ, μάλιστα, είναι υπεύθυνος για τα θέματα αυτά. Είπατε ότι οι κανόνες διαφάνειας του ΩΣΑ δεν σας βοηθούν και πολύ. Πώς θα μπορούσατε να το αναπτύξετε κάπως αυτό το σχόλιο σας. Αναφερόμαι στον κατάλογο που έχει όσα για, για ε, offshore ε, χρηματοπιστωτικά κέντρα και κάποιες τέτοιες ε, εξωεδαφικές δικαιοδοσίες. Υπήρχαν κάποιες τέτοιες δικαιοδοσίες που υπήρχαν στο μαύρο κατάλογο, στη μαύρη λίστα. Ε, λίγη όμως αυτή η μαύρη λίστα και στην γκρίζα λίστα δεν υπάρχουν και πολλά πολλά, δεν έχουν απομείνει και πολλοί, γιατί μερικές φορές για να φύγει κάποιος από τη μαύρη λίστα αρκούσε να υπογράψει κάποιες συμφωνίες. Αυτό εννοούσα όταν είπα προηγουμένω ότι τα θέματα αυτά του ΩΣΑ δεν μας βοηθούν και πολύ. Η κυρία Στίφλερ, αν θέλει το λόγο για να ολοκληρώσει. Ευχαριστώ. Θα ενημερώσω τον ε, εισηγητή, τον κύριο Πρέντα, για τα σχόλια και τις προτάσεις. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Να σας υπενθυμίσω τότε ότι η προθεσμία για τις ε, τροπολογίες λήγει στις 4 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, ενώ η ψηφοφορία θα γίνει στις 30 Σεπτεμβρίου. Το σημείο είναι έτσι ημερήσια διάταξη ε, με θέμα της πληροφορία που συνοδεύουν τι μεταφορέ χρηματοπιστωτικών χρηματικών ποσών αναβάλλεται για τις 16 ε, και 17 Σεπτεμβρίου, γιατί όπως σας είπα στην αρχή ο κύριος Δέβα απουσιάζει. Και περνάμε στο σημείο 10 για το Γενικό Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014. Όλα τα τμήματα. Ο εισηγητής μας, ο κύριος Κόρτες Λάστρα, έχει εκπονήσει πολλέ τροπολογίε για το Γενικό προπολογισμό και μάλιστα και άλλοι συνάδελφοι συνέβαλα με τι δικέ του τροπολογίε προκειμένου να ξεκινήσουν ή να παραταθούν πιλωτικά προγράμματα και σχέδια ή προπαρασκευαστικέ δράσει. Δυστυχώ, και ο κύριο Κόρτε Λάστρα απουσιάζει, κολλείεται και εκείνο και ζήτησε από τον κύριο Μπέργκμαν να τον αντικαταστήσει. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Μπέργκμαν για να μα παρουσιάσει τι τροπολογίε του εισηγητού, του κύριου Λάστρα και ενδεχομένω και κάποια άλλα χρήσιμα σχόλια για το σημείο 10. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τι έγινε με το 9, λέει ο κύριος Μίτσελ. Το περάσαμε. Είπα ότι αναβλήθηκε το σημείο 9 λόγω απουσίας του εισηγητού του κυρίου Ντέβα. Μας παρακάλεσε λοιπόν να αναβάλουμε το σημείο αυτό. Α, και η κυρία Γιώστρομ με απουσιάζει και μου ζήτησε να την εκπροσωπήσω εγώ. Μην ανησυχείτε, αναβάλλεται για τις 16-17 Σεπτεμβρίου το θέμα αυτό. Οπότε να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Μπέργμαν για να μας παρουσιάσει τις τροπολογίες του κυρίου Λάστρα για το Γενικό Προϋπολογισμό του 2014. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα διαβάσω το κείμενο που κατάρτισε ο κύριος Λάστρα και ελπίζω να γίνει αντιληπτό. Λέει λοιπόν ο Ρικάρδο. Συνάδελφοι, ζούμε εποχές λιτότητας Οπότε αναμένονται περικοπές από όλους, ακόμη και στα θέματα ανάπτυξης. Το θέμα με την ανάπτυξη είναι ότι τα κονδύλια που εξετάζουμε δεν είναι δικά μας. Είναι κονδύλια συνεργασίας και συνδρομής τους μειονεκτούντε για βασικά θέματα όπως είναι υγεία, εκπαίδευση, τροφή, είδωρ. Είναι θέματα που απειλούν την επιβίωση συνανθρώπων μας, γιατί ε, οι άνθρωποι αυτοί σε δυσμενεί συνθήκες δίνουν τον αγώνα της ζωής του. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε σε αυτού του ανθρώπου ε, ότι θα περικόψουμε τα κονδύλια της ανάπτυξη. Παρόλο που χώρες όπως ε, η Ολλανδία κάνουν δραστικέ περικοπές και σε αναπτυξιακά θέματα και λυπούμε ειλικρινά. Ελπίζω να επανέλθουμε στις αρχικέ προτάσει. Τον Ιούνιο στην Επιτροπή μας σχολιάσαμε τα θέματα αυτά στον τριμερή διάλογο και τα κράτη-μέλη ανέλαβαν τη δέσμευση να ενισχύσουν και να μην περικόψουν την αναπτυξιακή βοήθεια. Το Κοινοβούλιο δήλωσε ότι η οικονομική κρίση δεν είναι πρόσχημα για τη μείωση των δεσμεύσεών μας σε θέματα ανάπτυξης. Στον ανεξάρτητο όμως κόσμο που ζούμε, ε, είναι προ όφελό μα να ενισχύσουμε την ανάπτυξη, παρόλο που δυστυχώ υιοθετούμε συνταλτική ερμηνεία για αυτό το συμφέρον τη ανάπτυξη. Πρέπει να συνδράμουμε συνανθρώπου μα που ζουν σε πολύ χειρότερε ε, συνθήκε από ότι εμεί. Αυτό απαιτούν οι αρχέ μα και οι αξίε μα. Αυτό το θέμα αυτό δεν αφορά μόνο την Επιτροπή Ανάπτυξη. Τα μηνύματα αυτά θα πρέπει να τα προωθούμε προ όλε τι κατευθύνσει για να κρατήσουμε αλόβητου του προπολογισμού ανάπτυξη και ανθρωπιστική βοήθεια. Βέβαια, θα πρέπει να σχολιάσουμε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου για τον προπολογισμό του 2014. Θα πρέπει να ασκήσουμε ε, πιέσεις ώστε στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο, στο το όριο για τις εξωτερικές δράσεις, που είναι λιγότερο από το κατά 9% σε σχέση με το 2013, να το υποστηρίξουμε ή να αντισταθούμε στις ε, πιέσεις ε, για περικοπές, ενώ είναι αδύνατο σχεδόν να κρατήσουμε το επίπεδο του 2013. Πώς θα ελεγχιστοποιήσουμε τις περικοπές ε, σε ανάπτυξη και ανθρωπιστική βοήθεια. Ίσως θα πρέπει να, δώσουμε, να δείξουμε μεγαλύτερη ετοιμότητα από ό,τι αφέτ και να προγραμματίσουμε εμείς κάποιες περικοπές μαζί με εκπροσώπους των ε, πολιτικών ομάδων καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι καλό θα ήταν να επανέλθουμε στις πιστώσεις, επίπεδο πιστώσεων το 2013. Και αυτό ζητούμε στις τροπολογίες μας. Και η επαναφορά στα επίπεδα του 2013 φαίνεται ότι θα είναι η έκβαση και των ψηφοφοριών και σε εμά και στην ΑΦΕΤ, ώστε να ενισχυθεί ουσιαστικά η θέση της Επιτροπής προπολογισμού ότι φορά την ε, υιοθέτηση της ε, θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μάλιστα είναι πολύ σημαντικό ε, όλοι οι συνάδελφοι να αξιοποιήσουν τις εποφέ τους και να, προσπαθούμε, να, συνενο... να προσπαθήσουμε να συνεννοηθούμε με τα μέλη της Επιτροπής Προπολογισμών. Θα πρέπει να συντονιστούμε και με την Επιτροπή ΑΦΕΤ. Γιατί παρόλο που το ανώτατο όριο του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου για τις αναλήψεις υποχρεώσεων δημιουργεί αντιπαλότητα μεταξύ των επιτροπών ΑΦΕΤ και ΝΤΕΒΕ, κάτι που είναι αναπόφευκτο. Δεν υπάρχει όμως ανώτατο όριο για τις πιστώσεις πληρωμών. Υπάρχει μόνο για τις αναλήψεις υποχρεώσεων. Και το, ε, το ανώτατο όριο του πολιτού δημονομικού πλαισίου, που είναι πολύ χαμηλό, δυστυχώ έχει για ολόκληρο τον προπολογισμό. Τώρα, οι τροπολογίε δεν αφορούν μόνο ποσά, αλλά και τι παρατηρήσει και την κατανομή των δημοσιονομικών γραμμών γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μερικέ φορέ θέλει να συγχωνεύσει μερικέ δημοσιονομικέ γραμμέ χάρη ε, ε, ευελιξία και ελαστικότητα. Ει βάρο όμω τη διαφάνεια. Θα πρέπει να μπορούμε καλύτερα να στοχοθετούμε και να παρακολουθούμε τι δαπάνε. Γιατί αυτή τη χρονιά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνδύασε τι ε, συγχωνεύσει με, τη γεωγραφική κατανομή προβλέποντας υποκατηγορίες. Ε, διαφωνούμε με την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλουμε να παραφορά του δικτύου του επίπεδου του του 2013, γιατί με τη νέα κατανομή ε, καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την επαναφορά στο ποσό του 2013. Εμείς δεν θέλουμε να διπλασιάσουμε τις προηγούμενες δημοσιονομικές γραμμές και θα είναι δύσκολο να ασχοληθούμε και τα θέματα διακυβέρνηση ξεχωριστά γιατί τα θέματα αυτά αποτελούν απόσπαστο τμήμα των προκλήσεών μας και των σχεδίων μας σε συγκεκριμένο τομέα. Είτε αφορά την υγεία, την εκπαίδευση, τους μικροκαλλιεργητές, τις υποδομές ή οποιοδήποτε άλλο τομέα. Επίσης, εξαιτία ε, της παράτασης των διαπραγματεύσεων για το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και την ε, καθυστερημένη παρουσίαση του προϋπολογισμού, θα πρέπει ε, εντάχει να καταρτήσουμε τις τροπολογίες. Επίση έγινε μια αναπροσαρμογή των γραμμών απαράδεκτη στην πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ζητούμε, πολλές φορές ζητούμε πολύ περίπλοκες τροποποίησεις και πολύ τεχνικές προκειμένου να επανέλθουμε στο επίπεδο του 2013. Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν υπέβαλε την πρόταση της για την ανασυγκρότηση των δημοσιονομικών γραμμών έγκαιρα γιατί έτσι πολύ πολύτιμο χρόνο ε, για να υποβάλουμε πιο έγκυρες παρατηρήσεις. Και βρεθήκαμε σε μειονεκτική θέση. Δυστυχώς τα θέματα είναι πολύ ενδιαφέροντα και πολύ σημαντικά, ενώ δεν είχαμε αρκετό χρόνο για να τα αναπτύξουμε. Πάντως, ε, ο εισηγητής ε, Λάστρα προσβλέψει συνεργασία με τους συναδέλφους προκειμένου να διατηρήσουμε και στον προπολογισμό του 2014 λόγια τα κονδύλια για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Γκέρεντς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πούμε κάτι το οποίο να, να και να έχει συνέχεια σχέση με αυτό τον προπολογισμό. το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι το Συμβούλιο ε, σήκωσε τα χέρια. Δεν ανταποκρίνεται αυτή την πρόκληση. Και το Κοινοβούλιο επίση σε σχέση με αυτά που έλεγε στην αρχή τη ε, συζήτησης. Οπότε, για να μπορέσουμε να πούμε κάτι το ξεκάθαρο, θα πρέπει να δούμε το ότι θα ε, πρέπει να δούμε ότι θα πρέπει στα πλαίσια της CFP να λυθεί μια απόψη. Οπότε, σε σχέση με αυτά τα οποία μας είπε ο Τάις Μπέρμαν, είναι ότι θα πρέπει τελικά να κρυφθούν όλα την ώρα Αυτό λέει η λογική. Πάντως, για να διευκολύνουμε την επιλογή και για να μην χάνουμε το χρόνο μας, θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας διευκρινίσει κάτι. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων που τελούνται ε, μεταξύ Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής στο πλαίσιο του λόγου για ε, το CFP υπάρχει αυτή η διεκδίκηση του Κοινοβουλίου για περισσότερη ευελιξία. Τελικά, τι θα πει ε, ευελιξία που θέλει να αποσπάσει το Δηλαδή μήπως είναι έτσι οδηγηθούμε σε καλύτερη αξιοποίηση των πόρων για την πολιτική αυτή, για την ε, ελευθερική την σύρτη, Δηλαδή κατά πόσον μπορούμε με ένα τέτοιο εργαλείο να κάνουμε αυτό το οποίο θέλει να διεκδικήσει το Κοινοβούλιο. Και έτσι να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε κάπως περισσότερο ή σε αυτό το επίπεδο των εκταμιεύσεων που είχαμε το 2013 στα πλαίσια ε, το κάνουμε αυτό στα πλαίσια της χρήσης του προπολογισμού 2014. Γιατί δεν ξέρω αν το Κοινοβούλιο θέλει να εμπλακεί σε μια τέτοια ε, λογική του όλα ή τίποτα. Δεν το νομίζω πάντως εάν θέλουμε να δούμε τι επιχειρήματα υπάρχουν τόσο ώστε να μπορέσουμε να διευκολύνουμε την επιλογή των βουλευτών και να εξηγήσουμε συγκεκριμένα τι θα πει περισσότερη ευελιξία. Αυτό το έθεσα και στην τελευταία συνάντηση. Νομίζω ότι θα πρέπει να το ξανασυζητήσουμε επί τη βάση των ε, πληροφοριών που πρόκυψαν. Η πρόεδρος, ευχαριστώ. Μίτσο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο κύριο Κόρτε Λάστρα για την έκθεση και για τη δουλειά που έβαλε σε αυτή. Συμμερίζομαι την ε, αγανάκτησή του. Δεν ξέρω τι θα γίνει όταν θα φτάσει στη, στο τελικό στάδιο ψηφορία στο Κοινοβούλιο, εάν θα υπερασπιστούμε την άποψη ή τη γενική κατεύθυνση του εισηγητή στην Ολομέλεια. Εμείς μπορούμε να ελέγξουμε τι γίνεται εδώ σε αυτή την Επιτροπή και να στείλουμε ένα μήνυμα. Ένα όμως θα ήθελα να θίξω. Να αναφέρω ότι σε αυτούς τους ε, δύσκολους καιρούς, τους καιρούς ελιτότητας η σωστή και αποτελεσματική χρήση του προϋπολογισμού είναι το ό,τι σημαντικότερο. Γι' αυτό λοιπόν εξεπλάγει όταν είδα πώς κριτική άσκησε ο Βρετανός Πρωθυπουργό για τα διάφορα προγράμματα που έχουν σχέση με το νερό Και αυτό παρουσιάστηκε εχθέ ε, και στην Βουλή των Λόρδων στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία εξέφρασε τι ανησυχίε τη για το μέλλον των ε, ε, προγραμμάτων αυτών και τη εσπατάλη νερού που συμβαίνει. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα του νερού και της εσπατάλη του. Όταν λοιπόν ένας Υπουργό Εθνικού Κοινοβουλίου φτάνει σε τέτοιο σημείο ώστε να κάνει να εκφράζει δημόσια τις ανησυχίες τους είναι κάτι το οποίο πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη. Γι' αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε ίσως να μας ε, να αναφερθεί σε αυτές τις ε, ανησυχίες, να μας αναπτύξει τις απόψεις της, να μας πει πώς φροντίζουν να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διάθεση των πόρων. Να χρησιμοποιούμε δηλαδή τα κονδύλια μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στον κύριο Ιφτήλεμαν. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σημειώσει τις προτάσεις ε, και τις τροπολογίες στον προϋπολογισμό. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε την Επιτροπή για την πρόταση της ε, σε ορισμένων περικοπών του προϋπολογισμού και την εναρμόνιση του με, την, με το πρώτερο σχέδιο προϋπολογισμού. Αυτό έχει γίνει έτσι ώστε να φροντίσουμε να εξελιχθεί όσο το δυνατόν ομαλότερα η διάθεση των κονδυλίων. Υπάρχουν ορισμένα κριτήρια τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται για, τις, για ορισμένες υπηρεσίες και βασισμένοι σε αυτά θα δημιουργήσουμε ένα νομικό όργανο το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται ακόμα στα στάδια της υλοποίησης. Επίσης θα ακολουθήσουμε τα όσα προβλέπονται από το 21, άρθρο 21 κάθετος 02 του TCI όσον αφορά την ε, βιώσιμη ανάπτυξη και την ε, μείωση της φτώχειας από τη μία και την ε, καλή διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα από την άλλη, λειτουργούμε σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και φροντίζουμε να δημιουργήσουμε μία πρόταση που θα έχει επιμέρους συγκεκριμένες προτάσεις όσον αφορά την διάθεση των πονδυλίων του προϋπολογισμού. Όσον αφορά τώρα την νομενκλατούρα του προϋπολογισμού, εμείς θεωρούμε ότι η διανομή των κονδυλίων σε διάφορα αγαθά κοινή ωφέλεια, όπως έχει προταθεί από την Επιτροπή, θα είναι κάτι μη παραγωγικό. Να τονίσουμε επίσης το πόσο σημαντικό είναι να αποφύγουμε μια προσέγγιση κατά τομέα, διότι τα προηγούμενα προγράμματα έδειξαν ότι μια τέτοια ε, εφαρμογή έχει προβλήματα και τόσο στην εκτέλεση όσο και, στην, ε, και στον σχεδιασμό και επίσης μειωμένη αποδοτικότητα. Παρομοίως και με τις ε, γραμμές του προπολογισμού για την κοινωνία των πολιτών και τις τοπικές αρχές. Η πρώτερη εμπειρία μας έχει δείξει ότι ανάμεσα στην κοινωνία των πολιτών και στις τοπικές ε, αρχές ότι ο διαχωρισμός λοιπόν ανάμεσα αυτά τα δύο δημιουργεί προβλήματα. Επίσης, μία πρόταση, μία τροπολογία που έχει προταθεί να διατεθούν ορισμένα κονδύλια στο Αφγανιστάν. Εμείς θα θέλαμε να κρατήσουμε τον προϋπολογισμό για το Αφγανιστάν μαζί με τον γενικότερο προϋπολογισμό για την Ασία και όχι ξεχωριστά όπως έχει προταθεί. Ευχαριστώ. Δεν θέλει άλλο κανείς το λόγο. Ο κύριος Μπέρμαν, Εκ μέρους του Ρικάρντο θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για τα σχόλιά σας. Θα τα διαβιβάσω, θα τα λάβει υπόψη και να πω στου συναδέλφους ότι ε, ναι, μεν έχουμε απογοητευτεί από την πρόταση του προπολογισμού, αλλά ουσιαστικά έχουμε ένα πάγωμα του αναπτυξιακού προπολογισμού, κάτι που είναι το μη χείρον. Θα μπορούσαν να είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα, να είχαμε περικοπές αντί για πάγωμα. Ο, όλοι μας θα μπορούσαμε να καταψηφίσουμε τον προπολογισμό, γιατί παραμελούνται τα δικά μας προσφυλή θέματα, αλλά έτσι θα μέναμε χωρίς προπολογισμό. αν ο καθένας καταψήφιζε επειδή δεν είναι ικανοποιημένος. Ο κύριος Γκέρενς. Είπα προηγουμένως ότι θα ήθελα να ξαναθέσω μία ερώτηση που είχα αναφέρει και στο παρελθόν. Θα μπορούσαμε να έχουμε έστω και κάποιες γενικές ενδείξεις για την προστιθέμενη αξία που θα έχει η επιπλέον ελαστικότητα, η επιπλέον ευελιξία που δέχτηκε τελικά το Συμβούλιο στα πλαίσια του ημέρου διαλόγου ποιο θα είναι το πλεονέκτημα αυτής της ε, επιπλέον ευελιξίας. Αν δεν ευκαιρείτε να μας ε, δώσετε τέτοιες ενδείξεις προφορικά σήμερα, δεχόμαστε και γραπτός της εξηγήσεις σας. Πολύ ευχαριστώ. Κύριε σας. θα στείλουμε γραπτός απάντηση. Ωραία. Θα ψηφίσουμε τις τροπολογίες το απόγευμα. Ε, ολοκληρώσαμε την πρωινή συνεδρίαση λίγο νωρίτερα από το προβλεπόμενο, γιατί δεν ήμασταν και πάρα πολύ. Να σας υπενθυμίσω ότι η επανάληψη των εργασιών θα γίνει στις 3 στην ίδια αίθουσα. Καλό σας μεσημέρι.